Θεωρούμε ότι εφόσον δεν υπάρχει αντίληψη για το εκδοτικό, εγκρίνεται. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Γένσεν και Χόλμαγερ. Ψηφοφορία για τον προπολογισμό. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Votazione. Πέρας. Εγκρίνεται. Εάν θέλει το Συμβούλιο μπορεί να παρέμβει. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα συγχαρώ για την ψήφιση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημοσιονομικό έτος 2014. Το Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονό ότι το Ευρωκοινοβούλιο επιβεβαίωσε την συμφωνία που επετέφθη στην Επιτροπή Συνδιαλλαγή στι 11 και 12 Νοεμβρίου. Όπω όλοι θα γνωρίζετε, η συμφωνία περιλαμβάνει μια σειρά από κοινέ δηλώσει. Το Συμβούλιο στηρίζει ενθέρμως αυτές τις δηλώσεις και θα τιμήσει τις ε, τα σημεία που επετέφθη η συμφωνία. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αποτελεστώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών, τον κύριο Αλέν Λαμασούρ, και τους εισηγητές Αν Γένσεν, ε, Μόνικα Χολμάγκερ και Τζοβάνι Λαβία καθώς και τα άλλα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που συμμετείχαν στην ε, δημοσιονομική διαδικασία με πολύ επικοδομητική στάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα να διαβάσω ένα κείμενο, την κοινή δήλωση, βάσει τη οποία η Επιτροπή Συνδιαλλαγή επέτυχε συμφωνία στι 12 ε, Νοεμβρίου 2013. Ε, η συμφωνία αυτή κρίθηκε και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία η δημοσιονομική ε, εξελίχθη και βάσει των όσων ορίζουν οι συνθήκε και για το δημοσιονομικό έτος 2004 θεωρείται πέρα το φύσα. Ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσιονομικό έτος 2014 έχει τελεσίδικα εγκριθεί. Τον προπολογισμό θα συνυπογράψει θα υπογράψει μάλλον με σημερινή ημερομηνία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στην έκθεση ΔΕΑΝ. Κοινή ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λαβία. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φερνάντε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα βηματάκι πίσω, το Συμβούλιο θέλει να τοποθετηθεί για την έκθεση Λαβία. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μόλι μία τροπολόγηση για το διευθυντικό προπολογισμό υπερθυμών 9 για το 2014 από πλευρά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η τροπολογία αυτή συνάδει απολύτω με την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στην Επιτροπή Συνδιαλλαγή την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του κοινού κειμένου που αφορά τον προπολογισμό του 2014. Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του άρθρου 714 εδάφιο 4 γ για την συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να σα ε, βεβαιώσω ότι το Συμβούλιο εγκρίνει την τροπολογία αυτή, όπω ε, ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ό,τι αφορά τη θέση του Συμβουλίου για τον διευθυντικό προπολογισμό υπαριθμών 9 για το 2014. Άρα δεν χρειάζεται επιπλέον συνάντηση τη επιτροπή Συνδιαλλαγής όπως προβλέπεται από, άρθρο, από το άρθρο 314 εδάφιο 5 για τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έκθεση Μπέγκε. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μαρινέσκου. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μορέιρα. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Προύστ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση κλαίς. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση σαρτόρι. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φανίστε Ρόι. Κρέλ. Κυρία Μπερές. Κυρία Πρόεδρε, έχω ήδη τοποθετηθεί για το θέμα αυτό στην Σύνοδο της Δευτέρας διαπιστώνω ότι η διάσκεψη των Πρόεδρων παραβίασε τα άρθρα 50, 156 και 163 ε, και βάσει των ε, κανόνων του εσωτερικού κανονισμού δεν μπορεί να γίνει σε δημοκρατικέ συνθήκε η ψηφοφορία. Λυπούμε γι' αυτό. Έκανα μια τελευταία προσπάθεια χθε το βράδυ, προτείνοντα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξ ονόματο τη Επιτροπή Απασχόληση να περιληφθεί μια προφορική τροπολογία που θα επέτρεπε στην Ολομέλεια να τοποθετηθεί, τοποθετηθεί υπέρ ενό Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα 25% τη πολιτική συνοχή. Δυστυχώ αυτό δεν έγινε δεκτό. Κυρία Φερέιρα. Κύριε Φερέιρα, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να επαναλάβω εξ ονόματο τη ομάδα μα ότι υποβάλαμε διάφορε προτάσει τροπολογιών για την έκθεση αυτή την ε, πρόταση κανονισμού για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και θεωρούμε απαράδεκτο ότι η διαδικασία που προβλέπει αυτή η ψηφοφορία δεν επιτρέπει ούτε καν να ψηφιστούν αυτέ οι τροπολογίε μα. Θεωρούμε ότι είναι αντιδημοκρατικό περιορισμό αυτό και παραβιάζει τα δικαιώματα των Ευρωβουλευτών. Ε, είναι παραβίαση του δικαιώματο να υποβληθούν τροπολογίε και να ψηφιστούν υπέρ ή κατά, αλλά πρέπει να ψηφιστούν. Ε, γι' αυτό ζητούμε έντονα να αναθεωρηθεί αυτή η διαδικασία και να επιτρέπεται η ψηφοφορία των τροπολογιών μα και σε αυτή την περίπτωση. Ιδάλω δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ε, εφόσον δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία και η ψήφιση των τροπολογιών μα. Καταγράφουμε τις τοποθετήσεις αυτές, όμως πρέπει να προχωρήσουμε σε κάθε περίπτωση στην ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, αλλά όπως θυμήσατε, η διάσκεψη των Πρόεδρων ήδη έλαβε θέση. Ο πρόεδρος Σούλτ επίσης αποσαφήνισε το θέμα στην έναρξη της Ολομέλειας. Οπότε, χωρίς περαιτέρω συζητήσει θα ψηφίσουμε. Ομάδα 1, μπλοκ 1. Τελευταία παρέμβαση, τελευταία παρέμβαση. Παρακαλώ. Κύριε Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ Θέλω να ζητήσω να αναθεωρηθεί αυτή η τοποθέτηση. Θέλω να προτείνω μία τροπολογία, την 21η, που μιλά για την ε, μακρονομική αιρεσιμότητα, η οποία ουσιαστικά επιβαρύνει χώρες για τα διαρθωτικά ταμεία ε, με παραβιάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τα διαρθωτικά ταμεία. Είναι απαράδεκτο αυτό και θα ήθελα να τοποθετηθώ με προφορική τροπολογία. Allora, le vostre... Κοιτάξτε, ε, τα αιτήματά σας είναι σαφή, έχουν ήδη όμως απαντηθεί τα θέματα που γίνεται. Παρακαλώ, θέλετε και εσείς το λόγο. Δεν ρωτήσατε αν είναι κανείς αντίθετο σε αυτή την προφορική ε, τροπολογία. Εμείς είμαστε και ελπίζω να μας δώσετε την ευκαιρία πριν ε, συνεχίσετε να απορρίψουμε την προφορική τροπολογία της κυρίας Μπερές. Νόμιζα ότι το διευκρίνησα. Η τροπολογία θεωρείται μία αποδεκτή. Πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε το μπλοκ υπαριθμών 1 και μετά θα προχωρήσουμε στις τροπολογίες. Αυτό διευκρινίστηκε και στη διάσκεψη των Προέδρων και απήντησε ο κύριος Σούλτ την Δευτέρα. Θέτω λοιπόν σε ψηφοφορία το μπλοκ υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 489. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 480 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μωρά Σαρτιέ. Μπλοκ 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένα λεπτάκι. Εγκρίνατε. Κυρία Χάρμς, παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να πω ότι είναι σκανδαλώδες ε, ε, αυτό που γίνεται, ο τρόπος με τον οποίο ε, διευθύνεται τη συζήτηση. Η δική μου πολιτική ομάδα προσπάθησε, αποπειράθηκε να κάνει προφορική τροπολογία, το αρνηθήκατε και ξαφνικά επιτρέψατε στην κυρία Μπερές να κάνει προφορική τροπολογία. Εάν το δεχτήκατε αυτό πρέπει να δεχτείτε και τη δική μα παρακαλώ. Μα, ε, το γεγονό ότι παρουσιάστηκε. Κάποιο λέει ότι ε, απεσύρθη. Μα τι είναι αυτά που κάνετε, είναι τελείω αυθαίρετα. Κυρία Χάρμ, περιορίστηκα στο να ακολουθήσω όσα προβλέπει το καταστατικό. Εάν το θεωρείτε σκανδαλώδες, τι να σας πω, πρέπει να σεβαστούμε όμως και τους κανόνες επανερχόμαστε στην έκθεση Μωράν Σαρτιέ, πρόταση της Επιτροπής Ονομαστική Ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Όλμπριχτ. Μπλοκ 1. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Πακαρίναν. Βλόκ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψηφισμά. νομοστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μποστινάρου. Ε, μπλοκ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ 2 υπέρ με συγχωρείτε, όχι. Απευθεία πρόταση τη Επιτροπή. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Έκθεση Τζέλερ. Μπλοκ 1 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές με συγχωρείτε αποχές ε, εγκρίνεται. Το μαθηκό ψηφίσμα ονομαστική ψηφοφορία έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ρέγνερ Κράτσα. Άρχε, ε, ε, μπλοκ, μπλοκ ψηφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 33. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 50. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχετη ψυχοφορία, ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 68 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 83 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 48. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 84. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 καταπίπτει. 48 ονομαστική πληροφορία. Ε, ε, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 55-57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. πέρα. Εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέρας. Απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 ονομαστική άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Με συγχωρείτε. Ονομαστική ή άρχεται ψηφορία. πέρα. Απορρίπτεται. 79 ονομαστική ψηφορία. άρκετη ψηφορία. πέρα. Απορρίπτεται. 39 ονομαστική. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 67 ονομαστική. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 80 ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 81. Ονομαστική. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82. Ονομαστική. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθε... Συγχαρητήρια. Έκθεση Μπερές. Τροπολογία 1. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ε- Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκτο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έβδομο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Όγδο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. το τμήμα. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δέκατο τμήμα. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά, αποχές, έλεγχος, πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1, πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το τρίτο καταπίπτει. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Μπερέ, θέλετε το λόγο πριν την ψήφιση. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να είμαστε εδώ ότι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για να ολοκληρωθεί το νομοθέτημα αυτό και η πορεία του. Ήθελα λοιπόν να μα εξουσιοδοτήσετε να αναπέμψουμε το κείμενο στην Επιτροπή προ διαπραγμάτευση. quindi... Εντάξει. Θέτω λοιπόν σε ψηφοφορία την πρόταση τη εισηγητρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Λαβία. Τροπολογία 1. Με συγχωρείτε. Κύριε Ντεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρόκειται να ξεκινήσει η ψηφοφορία για τα πέντε νομοθετικά ε, ζητήματα που αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι πέντε ντοσιέ που ήταν πολύ κοπιαστικά στην εκτάσή του. Εργαστήκαμε δυόμιση χρόνια και περισσότεροι από 27 συνάδελφοι ε, ασχολήθηκαν από κοινού με τις διαπραγματεύσει για αυτό το σημαντικότατο αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν κέρια σημασία όλοι να υποστηρίξουμε τι συμβαστικέ λύσει με υπερψήφιση, ώστε να μην μην διακυβευθεί το σημαντικότατο έργο αυτής της τελευταίας δυόμισα αιτίας. Ευχαριστούμε κύριε Ντεκάστρο. Έκθεση Λαβία Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρασε, Εγκρίνεται. Έκθεση Καπόλα Σάντου. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρασε, Εγκρίνεται. Πρόταση τη Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική ψηφορία, άρχεται ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Νταντά. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καπόλα Σάντους. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, η μονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση DES. Μπλοκ 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπλοκ 2 καταπληκτή Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Βλάζακ. Τροπολογία 5. Υπέρ. Ο εισηγητής. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Βλάζακ. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα ψηφίσουμε την νομοθετική έκθεση που θα επιτρέψει σε δύο κράτη-μέλη ε, να έχουν διαρθωτικά ταμεία για ένα χρόνο ακόμα. Έγινε μια τέτοια συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η πλειοψηφία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης απλούστατα ε, ενέκρινε τη συμφωνία ενώ η Επιτροπή Προπολογισμών είχε ορίσει ότι θα πρέπει όλες οι χώρες να έχουν περισσότερο χρόνο, όχι μόνο δύο, για να μην γίνονται διακρίσεις. Κατά τα άλλα, ακόμα και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου θεωρεί ότι είναι προβληματική αυτή η τροποποίηση, ακριβώς διότι δεν δέχεται την αρχή της ίση μεταχείρισης όλων των κρατών μελών. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι εισηγητή, εγώ έκανα το καθήκον μου ε, και ε, έκανα τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο για αυτά που ήθαν οι συνάδελφοι ε, παρόλο που προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βλαζάκ. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1-4 καταπίπτουν. Πρόταση τη Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Όλμπριχτ. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω... Δεν δουλεύει το μηχανήμα, οπότε παρακαλώ να έρθει ένας τεχνικός. Ναι, ναι, ναι, θα το κοιτάξω. Έκθεση Όλμπριχτ. Τροπολογία. Παρακαλώ. Ο κύριος Ταβάρες. Κυρία Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε υπέρ τη έκθεση του κ. Όλμπριχτ που προβλέπει κονδύλια για την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων στι ευρωπαϊκέ νέε. Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία κατά κύριο λόγο. Τα κονδύλια αυτά δεν προσφέρονται με τρόπο τεχνικό ορθό, διότι οι χώρε που υπάρχει λιγότερη ενεργία έχουν περισσότερα κονδύλια και μιλάμε για χώρε που βρίσκονται σε πρόγραμμα ε, τη Τρόικα. Ε, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την, σύγχρον, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και Εδώ λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τα συμφέροντα των νέων και να ψηφίσουμε με, τρέπο, με τρόπο που να ε, αντικατοπιστούν σωστά οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο, όχι αυτέ που δεν έχουν όμω δημοκρατική νομιμοποίηση και που δεν συνάδουν και με του τεχνικού μα κανόνε. Ωραία. Ψηφοφορία τώρα, τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τρία Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέσσερα Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέντε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Έξι. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Έξι. Επτά, συγγνώμη, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Οκτώ, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εννέα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρόταση της Επιτροπής. Υπέρ. Με συγχωρείτε κύριε Όλμπερ. Όχι, όχι, Λάμστρομ. Μια παράκληση έχω προς τις υπηρεσίες. Ο κανονισμός προβλέπει ονομαστική ψηφοφορία σε άκρο σημαντικές ψηφοφορίες. Καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι των Πρασινών έχουν πρόβλημα με την έκθεση. Αλλά δεν θα πρέπει κάθε υποπαράγραφος και υποψηφοφορία να θεωρείται σημαντική. Παρακαλώ τις υπηρεσίες να τα ελέγχουν όλα αυτά λίγο πιο σοβαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Περνάμε στην ψηφοφορία για την πρόταση τη Επιτροπή. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Έκθεση Λέβιν. Έχει δικαίωμα να μιλήσει και να τοποθετηθεί η συγγήτρια. Δεν είναι στην αίθουσα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξή. Η έκθεση αυτή έχει συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή. Έγινε πάρα πολύ έντονη συζήτηση. Είμαστε κατά της πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή. Τελικά όμως ε, θα λυθούν τα προβλήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κυριμπάτι θα σεβαστούν αυτά που ισχύουν στον Ειρηνικό. Ευχαριστούμε. Τώρα ψηφίζουμε τη συμφωνία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκθεση Fox Hefner. Ο κύριος Hefner θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε τρεις προφορικές τροπολογίες τώρα στην ψηφοφορία. Θα ήθελα λίγο να σας εξηγήσω ε, πριν αρχίσει η ψηφοφορία για να μην χρειαστεί να διακόπτουμε. Είναι τρεις τεχνικής φύσεως τροπολογίες, οι δύο είναι και γλωσσικές μετά τα όσα ψηφίστηκαν στην Επιτροπή, ενώ η τρίτη σε συμφωνία με το συντάκτη της τροπολογίας θα βγάλει τη λέξη Βρυξέλλες για να διατηρηθεί η βασική χρειά της έκθεσης. Δεν μιλάμε για Βρυξέλλες Στρασβούργο. Αυτή την έκθεση μπορούν να την υπεψηφίσουν όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ανεξαρτήτως ε, της πεποίθησής τους για τις έδρες ή την έδρα του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στο εξή να αποφασίζει αυτόνομα και όχι ως υποτελές όργανο ε, της Ευρωπαϊκή κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Okay, grazie. Ε, Ευχαριστούμε. Όταν θα φτάσουμε στις προφορικέ τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε. Παράγραφος 1, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 2 μάλλον. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Εάν υπάρχουν αντιρρήσει, α ευχαριστούν, αλλιώ να συνεχίσουμε. Πρέπει να σηκωθούν ορθοί τουλάχιστον 40 βουλευτέ. Δεν θα ψηφιστεί η προφορική τροπολογία λοιπόν. Προχωρούμε. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Θέλετε έλεγχο για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Υψώστε τα χέρια παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος. Τρίτο τμήμα. Υπέρ, ε, άρκη ψηφοφορία, πέρας. Ε, απορρίπτεται. Να σηκώνετε περισσότερα τα χέρια σας παρακαλώ. Προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις. Ναι, υπάρχουν, οπότε θα περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Α. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσει στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική D, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική ο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αιτιολογική F, Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική. Ο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σα ευχαριστώ.